So, dear colleagues, good afternoon. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό σας απόγευμα. Θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημέρα διάταξη που είναι σύντομη, διότι όπως γνωρίζετε είχε προβλεφθεί να έχουμε τον, τον νομισματικό διάλογο με τον κύριο Ντράγκη. Η συνεδρίασή όμως αυτή θα, η συνάντηση αυτή θα γίνει τον Ιούλιο, 9 Ιουλίου. Ε, γι' αυτό και η μέσα διάταξη ε, έχει μόνο ένα θέμα, κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Έχουμε και κάποιους προσκεκλημένους εδώ, του συνάδελφου του Ιάκοπ Φον Φάιτσέκερ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια επιτυχή διαθεσμική διαπραγμάτευση Ίσως να ακούσατε ότι στις 30 Μαΐου η ομάδα διαπραγμάτευση τη ΕΚΟΝ έφτασε σε πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της πρότασης ECN Plus και της σχετικής οδηγίας για την ενίσχυση του πλαισίου ανταγωνισμού μέσω μεγαλύτερων εξουσιών προς τις ε, εθνικές αρχές ανταγωνισμού υπάρχει για το πακέτο σχετικά με την λίνιανση το θέμα της ε, διασυνορικής συνεργασίας, της ε, μεταβατικής περίοδου. Ο Επίτροπος Φεστάγκερ, ο οποίος συμμετείχε σε όλους τους τριλόγους, ε, ζήτησε, μια αξιολόγηση για τη μεταφορά της οδηγίας. Αναμένουμε μια επίσημη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Ε, θα γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες για να ολοκληρωθεί το συμφωνημένο κείμενο. Η Κορεπέρ στι 20 Ιουνίου θα εγκρίνει το κείμενο και εμείς θα συζητήσουμε εκ νέου ε, αυτό το, αυτή την προσωρινή συμφωνία κάποια στιγμή στο μέλλον, το κορινό μέλλον. Ε, σημαντικός αυτός ο τρίλογος στον τομέα του ανταγωνισμού. Να συγχαρούμε λοιπόν τον κύριο Σβάμπ, τον εισηγητή και όλα τα μέλη της Ευρωευτικής Ομάδας και βεβαίως και την γραμματεία και τους πολιτικούς συμβούλους που συνεισέφεραν. Να περάσουμε τώρα στο μοναδικό σημείο της ημέρας διάταξης για σήμερα είναι η γνωμοδότηση σχέδιο γνωμοδότησης μάλλον εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, επί της πρώτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος στήριξης διαθροτικών μεταρρυθμίσεων καθώς και η προσαρμογή του γενικού του στόχου. Βεβαίως θα γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Ρέτζι είναι η καθήλυνα αρμόδια, παρότι εμείς ε, δεν συμφωνούμε και τόσο. Ε, εγώ είμαι εισηγητής ε, για το θέμα αυτό από τη δική μας ομάδα. Θα είμαι σύντομος, θα αναφερθώ, στη δική μας Επιτροπή εννοώ, θα αναφερθώ μόνο σε τρία σημεία. Καταρχήν καλό θα είναι να γίνει μια μικρή παρουσίαση για το τι ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιο είναι το αντικείμενο μάλλον. Αυτή η πρόταση αποτελεί μέρο του πακέτου του Δεκεμβρίου 2017 για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Θέλει να τροποποιήσει τον κανονισμό για το πρόγραμμα υποστήριξη των ταμείων για να αυξηθεί το οικονομικό κονδύλιο και να προσαρμόσουμε τον γενικό στόχο έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και την υποστήριξη προς χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη. Όπως ξέρετε, η πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι να υπάρξει μια αύξηση 80 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2019-2020. Ε, ε, Ήταν επιτυχές το πρόγραμμα αυτό έως τώρα. Έχουμε πολλά αιτήματα από κράτη-μέλη αυξανόμενη η ζήτηση πρόκειται βεβαίως για μια πρόταση αρχική τώρα προτείνεται ένα νέο εργαλείο το οποίο θα είναι πλήρες ε, ευρύτερα στο πακέτο της, ε, για την Ευρωπαϊκή την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οπότε αυτό που προτείνουμε εμείς στην νομοδότησή μας ε, σχετίζεται με αυτά τα δύο έτη της επιμέρους αυτής αύξησης ε, του προπολογισμού, αλλά περιλαμβάνονται και κάποιες έννοιες που πιστεύω πως είναι σημαντικές για το μέσο αυτό στην επόμενη θητεία. Γίνεται αναφορά βεβαίως στη συνθήκη και στους στόχους της Ένωσης, ε, ε, στοιχεία που υπήρχαν και στο σχετικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, καλό όμως είναι να το συμπεριλάβουμε και εδώ στο κείμενο. Αυτή είναι η βασική τροπολογία μου. Επικεντρωνόμαστε σε τρία στοιχεία στην τροπολογία αυτή. Πιστεύω ότι πρέπει να διευρύνουμε την έννοια ε, των ε, διαθροτικών μεταρρυθμίσεων έτσι ώστε να επικεντρωθούμε περισσότερο ε, δηλαδή όχι αποκλειστικά να ασχολούμαστε με μέσα μείωσης του κόστους αλλά χρειαζόμαστε και στοιχεία που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, ε, την κοινωνική συνοχή και που θα μπορούν να υποστηρίξουν βιώσιμη ανάπτυξη και βεβαίως και περιβαλλοντικός και κοινωνικός βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η διεύρυνση λοιπόν της έννοιας της, μετα... της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που αποτελεί μέρος της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων έχει σημασία. Έχει σημασία να αποτυπώνεται και σε αυτό εδώ το έγγραφο, σε αυτό εδώ το κείμενο. Ε, το δεύτερο τώρα στοιχείο είναι ότι βεβαίως το κονδύλι αυτό δεν πρέπει να προέλθει από άλλα κονδύλια, τα χρήματα πρέπει να από άλλα κονδύλια ε, των κοινωνικών ταμείων. Σε γενικές γραμμές ε, θεωρούμε ότι τα ε, εργαλεία που έχουν να κάνουν με την ΩΝΕ δεν πρέπει να προέρχονται τα, τα σχετικά κονδύλια από αναδιανομή, αλλά να προέρχεται από άλλους πόρους. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο είναι και πιο φιλόδοξο από την Κομισιόν και το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το συνολικό ποσό του, ε, του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου έτσι ώστε να μην χρηματοδοτούμε το ΟΝΕ από την, από την ΟΝΕ και σχετικά εργαλεία από την κοινωνική πολιτική και τούμπαλιν. Επίσης υπάρχει μια πρόταση όπου εξετάζουμε τη δυνατότητα ε, να υπάρξει πραγματογνωμοσύνη προς τα κράτη-μέλη ε, αλλά οι εμπειρογνώμονες αυτοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και πρέπει να επιλέγονται σε, με, με τη σύμφωνη γνώμη του επιλεγμένου κράτους μέλους. Όλα αυτά θα τα βρείτε και στο κείμενο και στα εκτιμώντας. Απλή λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, σύντομη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους κοιόδους από το ΕΛΚ. Ο ε, Ευχαριστώ. Η Βάνα Μάλετιτς είναι στην Κροατία. Μου ανέθεσε να την εκπροσωπήσω. Είναι σκιώδης η συγγήτριά μας. Όπως είπες σωστά, ο κανονισμός θεσπίστηκε για, για, το, για, για το πρόγραμμα στήριξης τον Μάιο του 2017 και το πρόγραμμα αυτό διαρκεί από το 2017 στο 2020 με 142 εκατομμύρια ευρώ ε, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αιτήματα από τα κράτη-μέλη για την αξιοποίηση χρηματοδοτικής αρρωγής από το πρόγραμμα υπερέβησαν τα διαθέσιμα κονδύλια, ήδη στη δεύτερη χρονιά της εφαρμογής του προγράμματος αποφασίστηκε ε, ο προπολογισμό του προγράμματος να αυξηθεί κατά 80 εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η τροποποίηση του κανονισμού. Η εξασφάλιση επαρκών διαθέσεων ε, κονδυλίων μέσω του ΕΦΣΙ και άλλων ταμείων και μέσων τόσο από την, ε, από την EIB και την EBRD. Ωστόσο, αν ταυτόχρονα δεν εφαρμοστούν διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις από τα κράτη-μέλη, πρόκειται για σπατάλη, διότι στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο δεν θα βοηθούν τα κράτη-μέλη να αναπτυχθούν, αλλά θα αναβάλουν ε, στο και σοβαρά προβλήματα. Ταυτόχρονα επενδύσεις και μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι σημαντικότατη προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη. Μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό οι διορθωτικέ μεταρρυθμίσει και το αντίστοιχο πρόγραμμα στήριξη να συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα για κάθε κράτο μέλο. Το πρόβλημα που συχνά ανακύπτει είναι ότι οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις απαιτούν και πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα και υποστήριξη από όλα τα τμήματα της κοινωνίας, καθώς και από το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό κατά την εφαρμογή ε, των διατάξεων του κανονισμού να εξασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνεται υπόψη από τα κράτη-μέλη και η τοπική και περιφερειακή διάσταση καθώς και κάθε, άλλο, ε, κάθε άλλη ομάδα συμφερόντων της κοινωνίας κατά την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Στόχος μας είναι η επιτυχής εφαρμογή ε, και όχι ε, η, στα λόγια εφαρμογή κάποιων μεταρρυθμίσεων που δεν θα αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το ερώτημα των κοινωνικών ταμείων για, την, για το πρόγραμμα στήριξη ε, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων επίση είναι πολύ σημαντικό. Εγώ χαιρετίζω την πρόταση τη Κομισιόν αυτά τα επιπλέον 80 εκατομμύρια να χρηματοδοτηθούν από το Μηχανισμό Ευελιξίας ο προϋπολογισμός του οποίου ε, ανέρχεται σε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ και προβλέπεται ακριβώς προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ε, ελλείψεις, ελλείμματα ε, με βάση τον ισχύοντα προϋπολογισμό. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε αύξηση της χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών και μια σειρά άλλων κριτηρίων θα πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση των ε, μεταρρυθμίσεων, ιδίω εκείνων που έχουν θετικά αποτελέσματα σε διάφορου τομεί και ε, ενισχύουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή. Η επιτυχής εφαρμογή λοιπόν του προγράμματος μπορεί να οδηγήσει και σε μια αξιολόγηση για την επόμενη φάση του προγράμματος σε κάθε κράτος μέλος. Και αυτό μπορεί να βοηθηθεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών, ώστε στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα success story για το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Πιστεύουμε στις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη και πιστεύουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ε, πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Άρα ε, χρειάζεται να υπάρχει αφοσίωση και προσήλωση από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη δράση. Δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη έχουν ήδη την πρωτοβουλία μεταρρυθμίσεων, το πρόγραμμα στήριξη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να ενθαρρύνονται επιπλέον εθνικέ προσπάθειε και όχι να υποκαθιστούν ε, να υποκαθιστά το πρόγραμμα τη υπάρχουσα προσπάθειας. Στόχος λοιπόν είναι να ενισχυθούν οι ικανότητε των κρατών μιλών προκειμένου να προετοιμάζουν και να εφαρμόζουν διαρθωτικέ μεταρρυθμίσεις κατόπιν αιτήματο του κράτου μέλου και ε, να καλύπτονται μια σειρά από τομείς πολιτικής. Συμφωνούμε λοιπόν ότι οι ανθεκτικές οικονομίε που θα βασίζονται σε οικονομικέ και κοινωνικέ δομέ που θα ε, ε, επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να απορροφούν κραδασμούς και να ε, ανακάμπτουν βοηθούν στην εξασφάλιση κοινωνικής συνοχή. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν που ενισχύουν την ανάπτυξη αποτελούν σωστό εργαλείο για μια τέτοια κατεύθυνση. Κάποιες επιμέρους διαφορές έχουμε Ωστόσο, ε, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει προσοχή αν θέλουμε να συνδυάσουμε αυτό το πρόγραμμα με την διευκόλυνση για τη σύγκληση, ε, ιδίω όσον αφορά την προετοιμασία χρόνων για την προσχώρησή του στην Ευρωζώνη. Κάτι τέτοιο θεωρούμε ότι μπορεί να, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και αθέμητα κίνητρα σε εθνικού πολιτικού ε, προκειμένου να συμφωνήσουν να προσχωρήσουν Ευρωζώνη με αντάλλαγμα κάποια χρηματοδότηση η οποία όμως δεν, είναι, ε, δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν η χάραξη της πολιτικής και των προγραμμάτων να βασιστεί σε μακροπρόθεσμες προοπτικές. Όσον αφορά την αύξηση του κονδυλίου πρέπει να αιτιολογηθεί με ε, αξιολόγηση εκ των υστέρων όσον αφορά την χρήση των ε, χρημάτων και των κονδυλίων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και κατά πόσο αυτά έχουν πράγματι αποφέρει πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Στόχος, μας, ε, στόχος της γνωμοδότησής μας θα, πρέπει να είναι να συμπληρώσει την έκθεση που θα συντάξει η Επιτροπή Ρέτζι μέσω των τροπολογιών μας. Grazie, uh, ο κύριος Τρεμόζα για τους φιλελευθέρους. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, σήμερα το απόγευμα είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και να πάρω το λόγο για αυτό το θέμα, διότι είμαι τη γνώμη ότι το βασικό πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ελλειπή υλοποίηση του ενωσιακού δικαίου. Μέρο αυτού του προβλήματο είναι και αυτό ο κανονισμό θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε το οικονομικό χαρτοφυλάκιο του προγράμματος διευθυντικών μεταρρυθμίσεων, διότι πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πετύχει το στόχο, τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν παρομοίως τις βέλτιστες πρακτικές που υποτίθεται ότι τους γνωστοποιούμε με τον κανονισμό μας. Και ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συχνά αναγκάζεται να κινήσει διαδικασίες παραβάσεων παραβάσει κατά των κρατών μελών και αυτό δημιουργεί ένα πνεύμα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω μια από τις χώρες που εφάρμοζε σωστά το δίκαιο της Ένωσης ήταν ε, το Ρωμανό Βασίλειο. Κρίμα που φεύγεται και η Νορβηγία. Έχουν υλοποιήσει σε πολλούς τομείς το ενωσιακό δίκαιο με επιτυχία κιόλα και επειδή έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Άρα νομίζω ότι εδώ ε, ουσιαστικά αγγίζουμε την καρδιά του προβλήματος με, το, με την ομοδότηση αυτή. Το θέμα είναι να διασυνδέσουμε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι απλώς για να δώσουμε τριτά στα κράτη-μέλη, αλλά να διευκολύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, όχι απλώς να χαρίζουμε χρήμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο κανονισμό, είναι σημαντική αυτή η κίνηση και σε περίπτωση που βρούμε μια κοινή λύση θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο που κάνουμε τη δουλειά μα. Υπό την έννοια ότι έχει και κάποιο νόημα και σεβασμό η δουλειά που κάνουμε. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να είναι μια ε, ένωση που απλώς εκτελούνται κάποιες ε, επιταγές ε, που έρχονται άνωθεν, αλλά μια συλλογή βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται και διάφορες χώρες κινούνται σε μια σύγκληση, όχι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και τώρα για ένα άρθρο που διάβασα σήμερα στον αγγλικό τύπο, που αναφέρεται ε, η δυνατότητα το ενωσιακό δίκαιο εξαιτία των οργισμένων Ιταλών και ε, των ε, μάλλον Γερμανών και των τεμπέλιδων Ιταλών να καταρρεύσει το σύστημα του ενωσιακού δικαίου. Δεν πηγαίνουμε στην καλύτερη δυνατή κατεύθυνση και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις να ε, εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη. να πηγαίνουμε προς την ένταξη και την σύγκληση και να εργαζόμαστε αρμονικά και όχι σε πνεύμα διχόνοιας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για τους πρασίνους. Ο κύριος Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Λέτε δηλαδή ότι και η Ισπανία θα πρέπει να είναι μια ένωση βελτιστών πρακτικών και όχι μια ένωση μεταφορών χρήματος. Τέλος πάντων, πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με τον εισηγητή που λέει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο συνολική άποψη του τι είναι η διευθυντική μεταρρύθμιση, διότι μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά οι πράσινοι υποστηρίζουν τις βαθύτατες διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Το οικονομικό μας σύστημα δημιουργεί ανισότητες και οικολογικό αποτύπωμα τέτοιο που θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά στην διάρθρωση του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε διευθυντική μεταρρύθμιση στον νησιακό λεξιλόγιο, έχει πολύ συγκεκριμένο νόημα. Μιλάμε για ιστορική αγορά, για άνοιγμα των συνόρων ε, για το εμπόριο, την μείωση τη κυβερνητική παρέμβαση και ούτω καθεξή. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι όντω πρέπει να δούμε πιο σφαιρικά το νόημα τη ε, μεταρρύθμιση. Γι' αυτό να περιμένετε κάποιε τροπολογίε από τη δική μα την ομάδα. Ε, Παρεμπιπτόντω, οι διευθυντικέ μεταρρυθμίσει. θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο σκέλος των δαπανών, στο τι κοστίζει δηλαδή το κάθε τι, αλλά και στην πλευρά του εισοδήματος, ε, στο τι πόρους μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Δηλαδή, η καταπολέμηση της, της ε, φοροδιαφυγής και φοροαπάτης είναι ήδη ένα σημαντικό σκέλος των μεταρρυθμίσεων. Ως προς την πρόθεσή σας, κύριε Σιτά, να χρησιμοποιήσετε τον, ε, το πρόγραμμα αυτό για να ε, βοηθήσουμε στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να επιδιώξετε, αλλά όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, τα γνωρίζετε ότι σε πολλές χώρες τα προγράμματα αυτά, τα συστήματα αυτά, τα συνδιαχειρίζονται οι αρχές με τους κοινωνικούς εταίρους. Δεν είναι λοιπόν στα χέρια του κράτους. Ίσως εδώ λοιπόν να μην μπορεί να βοηθήσει τόσο πολύ το πρόγραμμα και να μην δώσουμε την εντύπωση ότι μέσω αυτής της αφορμή θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας λειτουργούν στις διάφορες χώρες ως προς τη διαχείρισή του. Κάτι ακόμα που θέλουμε να διευκρινιστεί είναι ότι το πρόγραμμα για τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις δεν θα πρέπει να πλήξει το σύστημα εταιρικών σχέσεων της πολιτικής συνοχής, το να χρησιμοποιηθεί ως ε, πρόσχημα για να ε, παρακάμψουμε τις αρχές ελέγχου που ασχολούνται με την σωστή υλοποίηση της νομοθεσίας. Γενικότερα πάντως επιμένουμε ότι πρέπει η έγκαιρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων να γίνει μια προϋπόθεση για τη σωστή ενεργοποίηση και χρήση του προγράμματος ε, των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων. Η ανάληψη ευθύνης πρέπει να γίνει πιο ε, σημαντική ε, αλλά από τη μια και τα εθνικά κοινοβούλια, από την άλλη και οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνες και να συμμετέχουν. Διαρκώς ακούμε για το έλλειμμα δημοκρατίας στην ε, οικονομική μας διακυβέρνηση. Όμως βλέπουμε τι έγινε στη Γερμανία με την Ομοσπονδιακή Βουλή, μάλλον με, τις κυβερνήσεις να να πάνε, με την κυβέρνηση να πρέπει να πάει στην Ομοσπονδιακή Βουλή για να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις και να εγκριθούν. Αυτό είναι κάπως η εξαίρεση. Τα περισσότερα κάτι μέλη, τα εθνικά ή έστω τα περιφερειακά κοινοβούλια δεν συμμετέχουν σχεδόν καθόλου, για να μην πω καν ε, λαμβάνουν γνώση του τι συμβαίνει ε, στις ε, συνεννοήσεις του εθνικού επίπεδου με το ευρωπαϊκό. Εάν θέλετε λοιπόν να, προωθηθεί, να μην προωθηθεί κι άλλο ιδέα του ελλείμματος δημοκρατίας, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι αρμόδιες αρχές, αυτές που θα πρέπει να επιληφθούν του θέματος, ε, επιλαμβάνονται όντως. Ευχαριστούμε ο κύριος Βιέγκας από την ΚΟΕΚ. δεν είστε εδώ. Από την EFTD, επίσης από την ENF κανείς, κάποιος στη διαδικασία CATSTI, ωραία. Κάποια σύντομα σχόλια για όσα είπατε. Καταρχάς σας ευχαριστώ Ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες για τις συνεισφορές τους. Με όσα άκουσα, πράγματα που περίμενα. Είναι ένα θέμα ευαίσθητο για όλους. Είναι η βάση, ε, νομίζω, το πρώτο σχέδιο του κειμένου για να βρούμε συμβαστικές λύσεις και νομίζω... αν σκεφτώ όσα υπόθηκαν. Και Είπες ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να δώσει τα λάθος κίνητρα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κανένα κράτος για 80 δις, τα 200 που θα κατανεμηθούν τέλος πάντων, θα το πάρει διαφορετικά. Είναι μια μικρή συμβολή στη διοικητική διαχείριση. Δεν καταλαβαίνω πάντως ακριβώς τον κίνδυνο. Ε, αλήθεια, για μένα ίσως να δίνουμε κίνητρο για να έρθει κανείς στην Ευρωζώνη, αλλά δεν φαντάζομαι ότι τη μεγάλη διαφορά θα την κάνει αυτό το κονδύλι. Η διάσταση αυτή της διοικητικής προπαρασκευής και ετοιμασίας είναι θετικό στοιχείο και καλώς ε, περιλαμβάνεται Επίσης διευκρινίζουμε ότι δεν υποστηρίζουμε μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Γιατί ταυτόχρονα έχουμε και μια διάσταση νομισματικής ένωσης. Για όσους δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Αλλά δεν είναι και η μόνη διάσταση. Μιλάμε για ένα ευρύτερο σύνολο μέτρων στήριξης. Και βεβαίως όλα αυτά είναι βάση, γίνονται βάση αιτήματος για να έρθω και σε αυτά που ραμών. Βεβαίω, η εφαρμογή του νοσιακού δικαίου είναι θεμελιώδη σημασία, γι' αυτό έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το σύστημα των ποινών και προστήμων. Οι καλέ διοικητικέ δυνατότητε όμω βοηθούν στην εφαρμογή του νοσιακού δικαίου, όντω, αλλά βρισκόμαστε σε έναν χώρο όπου βάσω των, ε, βάσει των αρχών μα ε, ξεφεύγει το νοσιακό δικαίου. Οι οικονομικές πολιτικές είναι ακόμα εθνικέ. Ε, και το σύστημα ε, της ε, ε, απόδοσης των αρμοδιοτήτων τώρα διευθετείται οι μεταρρυθμίσεις αποφασίζονται στο εθνικό, επίπεδο, στο εθνικό επίπεδο στα πλαίσια του εξαμήνου και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει κάποιες συστάσεις, όχι όμως να εκδώσει κανονισμό στα πλαίσια μιας κοινή αρμοδιότητας. Μιλάμε λοιπόν ακριβώς για τη δυνατότητα σε ένα σύστημα που βασίζεται στην ανάληψη ευθύνη. Ε, το πώς θα κινηθούμε στις κοινέ αρμοδιότητες στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής είναι ένα άλλο θέμα, αλλά δεν μιλάμε για αυτό εδώ. Εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο, ένα μηχανισμό που ενεργοποιείται μετά από αίτημα κάποιου κράτου μέλους και σκοπό έχει να βελτιώσει τις διοικητικές δυνατότητες. για να ε, προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Στήριξη λοιπόν προς τις, προς τις εθνικές αρχές για τα διοικητικά και οικονομικά μέτρα που θέλουν ε, να εφαρμόσουν. Η δυνατότητα δηλαδή των κρατών μελών να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις κατόπιν ετήν. Το άρθρο του Handelsblatt πάντως δεν με βρίσκει σύμφωνο. Στέκεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο βελτιώνοντας τις πολιτικές μας και ολοκληρώνοντας την οικονομική και νομισματική μας ένωση. Αυτός ο μικρός κανονισμός είναι ένα ελάχιστο τμήμα αυτής της μεγάλης προσπάθειας. και των υπόλοιπων φιλόδοξων προτάσεων που βρίσκονται υπό συζήτηση. Βεβαίω, όταν ανέφερα τον Ευρωπαϊκό Πολιόνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δεν υποστήριζα ότι αυτό που λέτε για τους κοινωνικούς εταίρους, σωστά βέβαια είπατε, ότι οι διαθετικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται αντιληπτές από μια ευρύτερη έννοια. Το έδειξαν οι εμπειρίες μας των τελευταίων ετών. Και όλο αυτό το φάσμα θεμάτων που καλύπτονται πλέον από τον Ευρωπαϊκό Πυλόν Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα έπρεπε όλα αυτά να ενταχθούν στην δυνατότητα των κρατομελών να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. σε πλήρη σεβασμό βεβαίω του εθνικού συνταγματικού αρχιτεκτονήματο και εφόσον απαιτείται η εμπλοκή και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, αυτό να ε, προβλέπεται. Νομίζω αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση, οπότε σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Προσβλέπω στις τροπολογίες σας. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο να βρούμε λογικές συμβαστικές λύσεις, πρόγραμμα για την ε, γνωμοδότηση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, διότι η Ρέτζη σκοπεύει να ψηφίσει τη δική της έκθεση στις 25 Ιουνίου. 25 ή Ιούλιο. Αρχές Ιουλίου. 25. Αυτό σημαίνει, αυτό συμφώνησαν οι συντονιστές της Επιτροπής μας, ότι έχουμε πολύ Αυστηρή προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 5η, 5 το απόγευμα. Και θα πρέπει να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά για να μπορέσουμε να τις ψηφίσουμε, να τις ψηφίσουμε στις 18-19 Ιουνίου πριν ε, ψηφιστεί η έκθεση της Ρέτζη. Θα πρέπει λοιπόν λίγο να προσαρμοστούμε σε αυτό το αυστηρό πρόγραμμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ αυτήν την ε, εκτάκτος συντομότατη συνεδρίαση. Η επόμενη... ...18 και 19 Ιουνίου, όταν μεταξύ άλλων θα ψηφίσουμε για αυτό το κείμενο.